αναβληθεί το σημείο αυτό. Υπάρχει ένα θέμα διαδικαστικό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ναι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε Σούλς, ελπίζω η Προεδρία σας να θεωρήσει σημαντικό την προστασία των δικαιωμάτων της του Τιμοσέγκο. Η γυναίκα αυτή έχει ληφθεί σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα και τώρα έχει μεταφερθεί σε ένα πραγματικό γκούλακ για να εκτίσει μια ποινή ε, από, η οποία έχει προέρθει από δυσφημιστικές ε, ε, κατηγορίες. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κοινοβούλιο μας δεν μπορεί να μείνει αθρανές ενώπιον αυτής της κατάστασης. Θα πρέπει να αναλάβει δράση πριν υπάρξει δραματικός επίλογος. Γι' αυτό ακριβώς σας ζητώ κύριε Πρόεδρε, η πρώτη σας επίσκεψη με την επίσημη η ε, ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι προς την Γιούλια Τιμοσέκο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στη δήλωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν σε σχέση με το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας. Θα ήθελα να καλωσορίσω με μεγάλη χαρά ως πρώην συνάδελφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την κυρία Χέλεν Τόνικ Σμιτ. Έχετε το λόγο. Ε, καλώς ήρθατε κυρία Πρωθυπουργέ. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για, την, ε, για το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας. Έχετε το λόγο, κυρία Τόνικ Σμιτ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, ηγέτες των πολιτικών ομάδων, κυρίες και κύριοι βουλευτέ και μέλη της Επιτροπής. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που παρευρίσκομαι μπροστά σας σήμερα για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Δανικής Προεδρίας. Ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους της εποχής μας ο πρόεδρος, τσέχος πρόεδρος Βάτσλαβ Χάβελ είχε πει. Εδώ και 20 χρόνια η Ευρώπη δεν χωρίζεται πια στα δύο. Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα επιτρέψει πια στον εαυτό της να ξαναδιαιρεθεί, αλλά αντίθετα θα μας δώσει νέες πρωτοβουλίες για ακόμη περισσότερη αλληλεγγύη και συνεργασία. Ο Χάβελ ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η Ευρώπη. Πρόμαχος μεγάλος μαχητής της ελευθερίας και της εφευρετικότητας και υπέρμαχος της ε, δημοκρατίας. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο της ιστορίας μας είναι κοινή μας ευθύνη να εφαρμόσουμε τις πεπιθήσεις του Χάβελ στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε το δυναμικό δυνατότητε της Ευρώπης για μεγαλύτερη ειρήνη, ευκαιρίες, ελευθερία και ευημερία. Αυτό είναι, αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη τη στιγμή που αναλαμβάνει την Προεδρία η Δανία. Ήθελα να σας μιλήσω σήμερα ως Πρωθυπουργό της Δανίας αλλά και ως πρώην μέλος του μεγάλου και μοναδικού αυτού κοινοβουλίου. Κάθε μέρα στα πολιτικά μηχανοστάσια σας λαμβάνονται αποφάσεις που θέτουν του θεμελιώδης λήθους στην οικοδόμηση της Ένωσης. Όπως και άλλα κοινοβούλια υπάρχουν έντονες συζητήσεις και διαφορές όπως και θα έπρεπε αλλά το ειδικό χαρακτηριστικό αυτού του κοινοβουλίου είναι η δέσμευσή του για την Ευρώπη και τους πολίτες. Είστε κοινοβούλιο της Ευρώπης και για την Ευρώπη. Για μένα ήταν πολύ ικανοποιητική η συμμετοχή μου στη σημαντική σας εργασία. Ήταν για μένα τιμή που υπηρέτησα στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων και στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ως τμήμα του συμφώνου που οδήγησε στην συνθήκη της Λισαβόνας. Και η ιδιαίτερη χαρά για μένα ήταν ότι συνέβαλα και εγώ στις αλλαγές που ενίσχυσαν δικαίως τις δικαιοδοσίες του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τους επόμενους έξι μήνες ζητώ την στήριξή σας, συνεργασία και τη συνεργασία σας. Αυτό είναι ζωτικό αν θέλουμε να πετύχουμε πραγματική πρόοδο στο βαρύ μα φορτωμένο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, ανήκω σε μια γενιά που το 80 ήταν νεολαία. Για πολλούς ήταν εποχή σκληρή με υψηλή ανεργία και λίγες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους που υπέφεραν και από τις περικοπές τους προϋπολογισμούς της παιδείας. Ήταν η γενιά που λεγόταν no future στην Ευρώπη όμως βρήκαμε ένα δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον. Είδαμε ηγέτες με όραμα σαν τον Χάβελ και καθώς περνούσαν τα χρόνια η Ευρώπη πραγματοποίησε την ενιαία αγορά γκρέμισε το τείχος του Βερολίνου και επανένωσε τη Γερμανία οδήγησε στη συνθήκη του Μάστριχτ και πραγματοποίησε τη διεύρυνση. Από την, απεσιοδοξία ακολούθησε μία εποχή ανάπτυξης προόδου και αισιοδοξία. Αυτό είναι επίτευγμα που πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γιατί λίγες δεκαετίες πριν η Ευρώπη από ήπειρο διαιρέσεων και πολέμων κατέληξε σε μία ένωση 27 εθνών βασισμένη σε πνεύμα δημοκρατίας και ανοιχτής συνεργασίας. Δημιουργήσαμε ένα μοναδικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την κοινοτική μέθοδο, που μας επιτρέπει με ελευθερία και δικαιοσύνη να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να μειώνουμε την πολιτιστική ποικιλότητα, ποικιλομορφία. Και Ακρογωνίως λίθος αυτής, αυτού του οικοδομήματος είναι οι κοινέ αξίες της αλληλεγγύης, της συμμετοχής και της συνεργασίας. Για μας δεν είναι απλώς ιδέες αυτά, αλλά πρακτικές καθημερινές πραγματικότητες. Γι' αυτό οικοδομήσαμε Ευρώπη με ισχυρή κοινωνική διάσταση. Θέλουμε και την ευημερία και την αλληλεγγύη, γιατί ξέρουμε ότι στο σύγχρονο κόσμο Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Στον αιώνα μας, ακόμα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, η δικαιοσύνη και οι ευκαιρίες είναι συστατικά στοιχεία της αποτελεσματικότητας η οποία είναι η πηγή για σωστές επενδύσεις στο μέλλον και στη δικαιοσύνη. Αυτό το μείγμα είναι η βάση της ευρωπαϊκής επιτυχίας. Αυτό το τονίζω ιδιαίτερα σήμερα όχι για να αποτίσω φόρο τιμή στο παρελθόν αλλά για να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη για το μέλλον. Όλοι εδώ ξέρετε ότι η Ευρώπη ζει μια βαθιά οικονομική κρίση που έχει κλειδονίσει τα θεμέλια της συνεργασίας μας. Η ανάπτυξη είναι χαμηλή, το χρέος υψηλό και η ανεργία αυξάνεται. Η ανασφάλεια στην καθημερινή ζωή είναι μια πραγματικότητα για εκατομμύρια ευρωπαϊκών οικογενειών και λόγω της φύσης αυτών των προβλημάτων οι πολίτες της Ευρώπης ζουν συνεχώς μειώσεις και περικοπές. Αυτό την πρόκληση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά για να επανέλθει η εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, για να υπάρξουν νέα θεμέλια για την ανάπτυξη και την πρόοδο και για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού προτύπου. Αυτό το χρωστάμε σε όλες τις γενιές, σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα όμως στους νέους. Οι νέοι ζητούν κάτι που είναι απλώς λογικό και δίκαιο. Πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες μόρφωσης και απασχόλησης με τις προηγούμενες γενιές. Μια ευκαιρία δηλαδή να συμβάλλουν και αυτοί στην ανάπτυξη της κοινωνίας και σε ένα σίγουρο μέλλον. Θα κάνουν ό,τι μπορούν αλλά δεν θα το πετύχουν παρά μόνο αν τους ενθαρρύνουμε και τους το επιτρέψουμε. Αν θέλουμε και αυτοί να μας φροντίσουν στο μέλλον πρέπει και εμείς να τους φροντίσουμε από τώρα. Αυτό είναι το συμβόλαιο μεταξύ των γενεών και πρέπει να το τιμήσουμε. Πρέπει να επιδείξουμε την ίδια αποφασιστικότητα στην διαχείριση των οικονομικών μας. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό προπύργιο κατά της κοντόφθαλμης κερδοσκοπίας. Το μόνο μέλλον που μπορεί να έχουν οι κοινωνίες μας είναι αυξημένη ανταγωνιστικότητα και η βάση γι' αυτό είναι ότι η σταθερότητα δημιουργεί ανάπτυξη και καινοτομία. Οι περικοπές δεν είναι μείωση της αλληλεγγύης. Στις σημερινές συνθήκες είναι προϋπόθεση για την αλληλεγγύη. Είμαι βέβαιη Βέβαια λέγω ότι οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν αυτό. Αν εφαρμοστεί δίκαια, είναι έτοιμοι να κάνουν θυσίες, αλλά όχι και του εαυτού τους. Θα δεχτούν τη λιτότητα αν υπάρχει και δικαιοσύνη, αλλά θα αντισταθούν σε αυτήν αν είναι η λιτότητα άδικη. Ως Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να ανταποκριθούμε σε αυτή την πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, η μοίρα της Ευρώπης είναι η μοίρα της Δανίας. Αυτό το γνώριζε η Δανία για δεκαετίες. Πριν από 40 χρόνια ήταν τμήμα της πρώτης διεύρυνσης της κοινότητας και οι εταίροι μας τότε μας έδωσαν τον ίδιο πρώτο εκείνο χρόνο και την Προεδρία. Πριν από 30 χρόνια είχαμε την Προεδρία σε περίοδο του ψυχρού πολέμου και οικονομικής αβεβαιότητας αλλά και στην πρώτη περίοδο του εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 20 χρόνια πριν είχαμε την Προεδρία την εποχή που άρχιζε η ενιαία αγορά και πριν από 10 χρόνια είχαμε την Προεδρία τη στιγμή που η Ένωση τιμούσε την ιστορική της δέσμευση για την Ένωση της Ευρώπης. Ε, και τώρα πάλι αντιμετωπίζουμε μια κρίσιμη περίοδο. Τους επόμενους 6 μήνες θα κάνουμε και πάλι προσπάθεια να προωθήσουμε την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν από τους ηγέτες τους δράση και αυτό είναι σωστό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Η δημοκρατική πολιτική κρίνεται από τα αποτελέσματα, όχι από τις προθέσεις. Η Ιδανική Προεδρία α, θα κάνει ό,τι μπορεί τους επόμενους έξι μήνες για να διασφαλίσει ότι η Ένωση θα συνεχίσει να παράγει απτά αποτελέσματα και χρήσιμα που να ωφελούν όλους τους Ευρωπαίους ηλικιωμένους και νέους φοιτητές και εργαζόμενους στον Νότο και στη Βορρά. Οι προτεραιότητες μας είναι λοιπόν οι εξής. Πρώτον, η Δανική Προεδρία θα δημιουργήσει, θέλει να δημιουργήσει μια υπεύθυνη ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε από την κρίση η Ευρώπη να επανέλθει στην ευημερία και την ασφάλεια για όλους τους πολίτες. Πράγμα που απαιτεί πειθαρχία και πολιτική θέληση από όλους για να εφαρμόσουμε τους νέους κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης, governance. Χρειαζόμαστε έναν υπεύθυνο προϋπολογισμό και τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών. Δεύτερον, θα εργαστούμε για μια πιο δυναμική Ευρώπη η ανάπτυξη στην Ευρώπη πρέπει να επανέλθει και να είναι βιώσιμη. Πρέπει να προωθήσουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας τουλάχιστον για τους νέους. Ο εξυγχρονισμός και η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς είναι ένα κλειδί για αυτή την προσπάθεια και πρέπει να βοηθήσουμε τις εταιρείες μας να εκμεταλλευτούν όλες τις ευκαιρίες που έχουν σε συνεργασία με τις αναδυόμενες οικονομίες εκτός Ευρώπης. Τρίτον, θέλουμε να πρασινίσουμε την Ευρώπη. Η Ένωση έχει μία πολιτική για την ενέργεια και τα κλιματολογικά. Είμαστε από τους κύριους παίκτες στο παιχνίδι αυτό, αλλά για να διατηρήσουμε τη θέση μας και να ενθαρρύνουμε και τους άλλους χρειάζονται νέες πρωτοβουλίες για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Πάνω από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σχετίζονται με το περιβάλλον εδώ υπάρχει τεράστιο δυναμικό, τεράστιες δυνατότητες, αλλά υπάρχει και ο πραγματικός κίνδυνος η έρευνα για την υψηλή τεχνολογία να μετακινηθεί εκτός Ευρώπης. Η Δανική Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε η δημιουργία πρασίνων θέσεων εργασίας να παραμείνει στην Ευρώπη. Τέταρτον, θέλουμε μια ασφαλή Ευρώπη σε, ένα παγκοσμιοποιημένο, σε μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση μόνο μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσπάθεια θα είναι αποτελεσματική για να διασφαλίσει τις ελευθερίες και την ασφάλεια των πολιτών για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία και το διαμεθοριακό έγκλημα για να διαχειριστούμε καλύτερα τα σύνορά μας και για να λειτουργήσει ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και πέρα από μας η φωνή της Ένωσης πρέπει να ακουστεί ακόμη καθαρότερα για να προωθηθούν οι κοινέ μας αξίες και τα συμφέροντά μας. Η Προεδρία θα στηρίξει λοιπόν και την ύπατη εκπρόσωπο για την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Η δημοσιονομική πειθαρχία λοιπόν, η ανάπτυξη και οι θέσει απασχόλησης, η πράσινη πολιτική και η φωνή της Ευρώπης στο μέλλον για μια ασφαλέστερη Ευρώπη. Αυτά είναι οι προτεραιότητες μας. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι μέσα στην οικονομική κρίση, εν μέσω της οικονομικής κρίσης δεν αναμένω να είναι εύκολη η δουλειά της Δανικής Προεδρίας αλλά μπορώ να σας διασφαλίσω ότι η Προεδρία μας δεν θα πισωγυρίσει δεν είναι στο χαρακτήρα μας προφανώς μια Προεδρία δεν μπορεί από μόνη της να έχει αποτελέσματα χρειάζεται συνεργασία από όλους τους ενδιαφερόμενους τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά όργανα και την κοινωνία των πολιτών. Χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η δική σας βοήθεια και στήριξη στο Κοινοβούλιο θα είναι κάτι το ζωτικό στην προσπάθεια αυτή. Κυρίες και κύριοι, ως Πρωθυπουργό τη Δανία σήμερα σας διαβεβαιώνω ότι προσωπικά είμαι δεσμευμένη στην Ευρώπη είμαι Ευρωπαία και πάνω απ' όλα για τα παιδιά μου. Γιατί γνωρίζω ότι η ασφάλειά τους, οι ευκαιρίες τους, η ελευθερία τους θα εξαρτηθούν από την ασφάλεια, τις ευκαιρίες και την ελευθερία της προηγούμενης γενιάς. Η Ένωση είναι το καλύτερο εργαλείο για την ενδυνάμωση τέτοιων συνθήκων διαβίωσης και στην Ήπειρό μας και σε ολόκληρο τον κόσμο κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι. Το κυριότερο μέσο για την διασφάλιση των στόχων μας είναι αυτά που θα κάνουμε σε περιόδους κρίσης και όχι όταν τα πράγματα είναι όλα εντάξει. Όπως σας είπα ήδη, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι τρεις βασικά. Πρώτον, πρέπει να βασιστούμε στους κανόνες Λήψη των αποφάσεων που ήδη έχουν εγκριθεί στην Ένωση γιατί είμαστε Ένωση που βασίζεται στη συνεργασία και τη δημοκρατία. Σε περίοδους κρίσεων οπότε και πρέπει να ληφθούν σκληρές αποφάσεις και συμβιβασμοί το βασικό εργαλείο η κοινοτική μέθοδος είναι σημαντικότερη παρά ποτέ. Βασιζόμενοι λοιπόν στους βασικούς μας κανόνες και διαδικασίες δεν είναι κάτι που συμφέρει μόνο μικρά κράτη-μέλη όπως η Δανία. Είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ένωσής μας. Είναι αυτό που καθιστά τη συνεργασία μας τόσο ισχυρή και βιώσιμη. Και αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα είναι μέρος της λύσης στην κρίση και όχι του προβλήματος. Η έξοδος από την κρίση σημαίνει περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Τις παρούσες συνθήκες η εσωστρέφεια σημαίνει ότι δεν βλέπει κανείς την πραγματικότητα. Και καθήκον των ηγετών της Ευρώπης είναι να το δείξουν αυτό στους πολίτες και στον έξω κόσμο. Γιατί τα πρακτικά αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η Ευρώπη θα δημιουργήσουν περισσότερη εμπιστοσύνη. Τρίτον, πρέπει να βγούμε από την κρίση με απνέπαφες τις αξίες μας. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί είναι κάτι το σωτικό για να σταθεροποιήσουμε τις οικονομίες μας, αλλά όταν αφού μάλλον η οικονομική πτυχή της αγοράς μα, της αγοράς μας υπήρξε επιτυχία, πρέπει να παραμείνει σαν βασικό στοιχείο της δουλειάς μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δοκιμάζεται σκληρά η Ένωση από την κρίση. Οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν αναλάβει τεράστια ευθύνη για να διασφαλίσουν την οικονομική σταθερότητα στην περιοχή μας. Το λεγόμενο δημοσιονομικό συμβόλαιο θα παίξει ένα ρόλο κλειδί στη σταθεροποίηση του ευρώ και αυτό είναι συμφέρον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν πρέπει να μας παραπλανά η κρίση. Είναι πιο φανερό παρά ποτέ ότι είναι κοινή η μοίρα μας. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεργαστούμε. Αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε το όραμα του Βάτσλαβ Χάβελ για τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, πρέπει η Ευρώπη να ξαναρχίσει να λειτουργεί. Και μόνο μαζί θα το πετύχουμε. Σας κάτι ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι.